Uh, Μάλιστα. Καλημέρα σας. Ελπίζω να είναι όσοι χρειάζεται εδώ για την πρώτη έκθεση. Πρώτα θα εγκρίνουμε τη ημερήσια διάταξη. Δύσκολη αίθουσα, δεν σας βλέπω καλά όλους. Θα περιμένετε μέχρι να σας βλέπω. Λοιπόν, θα μετά την ψηφοφορία οι ανακοινώσει της Προέδρου για να έρθουν κι άλλοι. Άρα περνάμε στο 3 και 4. Συμφωνία συνεργασίας της Ένωσης για την πολιτική συνεργασία κλπ. κλπ. Ο εισηγητής είναι ο Γεώργιος Κούτας. Ευχαριστώ, Σάρων. Θα συζητήσουμε εδώ μαζί το 2 και το 3 γιατί συνδέονται. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποφασίσαμε να γίνει ένα ευρύτερο ψήφισμα για τις συμφωνίες συνεργασίας για την πολιτική ανταγωνισμού με βάση την τρέχουσα διαπραγμάτευση Ένωσης Ελβετίας δεύτερης γενεάς. Μια τέτοια συμφωνία με την Ελβετία είναι νομίζω απαραίτητη λόγω της στρατηγικής σημασίας της, Σουηδίας, της Ελβετίας για την Ένωση και πιστεύω ότι η τιμωρία των διαμεθοριακών παραβιάσεων του δικαίου θα είναι πιο αποτελεσματική αν αρχίσει να ισχύει αυτή η συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία αυτή δεν είναι δεσμευτική ως προς τη συνεργασία και αφήνει μεγάλο περιθώριο για τον ορισμό του ζωτικού συμφέροντος αναπερίπτωση ανάλογα με την αίτηση που θα έχει κάνει το α ή το β μέρος. Η καινοτομία αυτών του είδους συμφωνιών είναι η δυνατότητα της Κομισιόν και της ανάλογης επιτροπής της Ελβετίας να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι θετικό και πρότυπο για τις μελλοντικές τέτοιες συμφωνίες. Εκτός αυτού η Ένωση θα έπρεπε να εγκρίνει ένα γενικότερο πλαίσιο για, τις, ε, για την ελάχιστη κοινή βάση για οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα αλλά θα διαθέτει πάντοτε ένα περιθώριο ελιγμών ανάλογα με την περίπτωση. Βεβαίως πρέπει να καθοριστεί και ένας μηχανισμός για την ασφαλέστερη λειτουργία των ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, επίλυση διαφορών ιδιαίτερα αν χρειαστεί στο μέλλον να γίνει κάποια αποκάλυψη λόγω διώξεων. Δυστυχώς τελευταία στην αρμόδια επιτροπή The Swiss Parliament. του Κρατικού Συμβουλίου της Ελβετίας ε, από εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα ανησυχία ως προς το κατά πόσον θα είναι προστατευμένες οι εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εγκρίνει τη συμφωνία. Την έχουν παγώσει και αυτό είναι περίεργο γιατί αρχάς Νοεμβρίου είχα οργανώσει και εγώ μια ακροάση και συνεννοήθηκα και με τον Ελβετό πρέσβη εδώ Μπαλζεράτη και δεν προέβλεψε κανείς να υπάρξει πρόβλημα για την έγκριση της συμφωνίας από την Ελβετική Βουλή. Τώρα, η Κομισιόν εδώ είναι παρούσα και γι' αυτό ίσως καλύτερο είναι να τους ρωτήσουμε απευθείας τι περίπτωση υπάρχει να απορρίψει η Ευρωετική Βουλή αυτή τη συμφωνία ή να την εγκρίνει. Γιατί νομίζω θα έχουν περισσότερες πληροφορίες από μας. Προς το παρόν έχει συνταχθεί το ψήφισμα και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου γνωμοδότησε και γι' αυτό προτείνω να προχωρήσουμε. Αν η Ελβετική Βουλή αποφασίσει να την απορρίψει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά προς το παρόν προτείνω να συνεχίσουμε τη διαδικασία και να δούμε τι θα γίνει γενικότερα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ο Σκιώδης Μάρκος. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή. Μπορώ να συμφωνήσω με την ε, πρόταση ότι η πρόταση αυτή δεν είναι κάτι το ρηξικέλευθο, αλλά πάντως δημιουργεί ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή κατά τρόπο εμπιστευτικό, εμπιστευτικό ε, πληροφοριών για θέματα ανταγωνισμού. Πρέπει να φροντίσουμε να μην παραμείνει ένα blueprint, ούτε μία μπλε παύση για ε, τα θέματα αυτά τη συνεργασία στον ανταγωνισμό ή με την Ελβετία είναι κάτι το αρκετά σημαντικό. Πρέπει να το προωθήσουμε και να εξασφαλίσουμε συμβατότητα μεταξύ των δύο συστημάτων για την ε, πρόσβαση και την διάθεση πληροφοριών. Και πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει εν τέλει να υπερψηφίσουμε την ε, έκθεση. Είναι περιορισμένο το περιθώριο ε, δράσης νομικά. Έχετε διερμηνία στα αγγλικά τόση ώρα. Δεν έχετε στα αγγλικά. Κρίμα. Όχι, ήταν τα ακουστικά μου χαλασμένα, αλλά τα φτιάξα. Άρα δεν ήταν η διερμηνία, ήταν η ηλεκτρονική της μεταφορά μέχρι τα αυτιά σας. Καλώς, για να συνεχίσω λοιπόν στα γερμανικά, παραμένει ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού και στην ευρωπαϊκή στη σχέση με τρίτα κράτη παραμένει ένα μαύρο κουτί, πράγμα για το οποίο βέβαια λυπούμε. Από την άλλη και όπως πόθηκε και νωρίτερα και λόγω των πολύ περιορισμένων δομών, διαδικασιών, ε, και διατυπώσεων είναι δυνατή η συνεργασία και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε εν τέλει να υπερψηφίσουμε την συμφωνία με δεδομένο ότι θα υπάρχει περιθώριο και στο μέλλον για περαιτέρω επεξεργασία της διευκρίνησης λεπτομεριών και βελτίωση της διαφάνειας. Ευχαριστώ. Νίλς Άλντερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. <laughs> Και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Είναι ένας νέος τύπος συμφωνίας. Συμφωνία δεύτερης γενναίας. Που ελπίζω ότι θα φέρει τα αποτελέσματα που μας υπόσχεται. Παγκοσμιοποιημένο ο κόσμο μα. η Ελβετία είναι στο κέντρο και πολύ κοντά σε εμά Ασφαλώ θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ο κύριο Κούτο λοιπόν έχει κάνει τι σωστέ επιλογές και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν βλέπω να είστε κανένα άλλο από το Σκιώδης, να είναι παρόν κανεί άλλο σκιώδη. Θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο του Κοινοβουλίου να λάβει τον λόγο. Όχι. Η Επιτροπή μήπω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και καταρχάς ευχαριστώ πολύ τον ε, εισηγητή και τους ε, λοιπούς βουλευτές για την ε, θαραλέα αντιμετώπιση του θέματος, όχι μόνο της συμφωνίας δηλαδή, αλλά και της γενικής πολιτικής που έχουμε στη διεθνή συνεργασία. Ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά λόγια και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, για τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Τα παρουσίασε ο κύριος ε, Κούτας. Όλο και πιο πολλές συγχωνεύσεις ε, είναι διεθνείς. Συνεργαζόμαστε με τις ελβετικές αρχές και γενικά με όλες τις αρχές που βρίσκονται άλλωστε στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας μας, ενημέρωσε ο κύριος Κούτας για τις ανταλλαγές των στοιχείων αυτών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μόνο όταν ε, διερευνούν ε, την ίδια ή παρόμοια ε, συμπεριφορά οι αρμόδιες αρχές και η ανταλλαγή θα γίνεται επί τη βάση αυτού μόνο. Στοιχεία που αφορούν ενδεχόμενη αμνηστία, ε, άφεση κτλ. δεν θα ανταλλάσσονται παρά μόνο αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών. Για την ερώτηση του κυρίου Κούτας αλλά και άλλων ε, βουλευτών για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης στην Ελβετία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η αρμόδια για την κύρωση της συμφωνίας ε, αρχή από πλευρά Ελβετικής, που είναι η Βουλή στην Ελβετία, έχει αναβάλει μέχρι τον Δεκέμβριο αρχικά, μετά μέχρι τον Ιανουάριο, την ε, συζήτηση και ψηφοφορία. Πίσω από αυτήν την επιλογή κρύβονται κάποιες μέρημνες που έχουν να κάνουν με την παράλληλη τροποποίηση του, ε, του εθνικού δικαίου περί ανταγωνισμού, του ελβετικού δηλαδή δικαίου και τη εισαγωγή σε αυτό ενδεχομένως της δυνατότητας για μια επιχείρηση να υποβάλει προσφυγή ή ένσταση σε ε, απόφαση της αρμόδιας αρχής για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο βέβαια μας ανησυχεί σε έναν βαθμό, εάν δοθεί αυτή η δυνατότητα για την ε, προσφυγή κατά τις αποφάσεως για την ανταλλαγή πληροφοριών και ενταχθεί τελικά στο εθνικό δίκαιο της Ελβετίας, θα είναι μάλλον δύσκολη ανταλλαγή πληροφοριών για μας. Ε, προκειμένου λοιπόν και χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο και τις επιλογές του Ελβετικού Κοινοβουλίου, αυτό που κάνουμε όμως είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε στις επαφές μας και με το ε, Ελβετικό Κοινοβούλιο και γενικά με τις Ελβετικές Αρχές για να τους εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτών των ανταλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς, τι είδους πληροφορίες διαθέτουμε και γενικά να προσπαθήσουμε να τους καθησυχάσουμε ως προς την συμφωνία αυτή. Δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε τι θα συμβεί εν τέλει. Η ελβετική κυβέρνηση, ωστόσο, οι ελβετικές αρχές είναι ιδιαίτερα ε, αποφασισμένες να προωθήσουν αυτή τη συμφωνία, όσο και εμείς άλλωστε, για να, και να πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν το ε, Κοινοβούλιο, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την διαδικασία αυτή της, αναθε... της ένστασης της προσφυγής. Επίσης, ένα επιχείρημα που έχουμε είναι ότι έχουμε το πιο ανεπτυγμένο δίκτυο αρχών ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και όπου πάλι δεν προβλέπεται προσφυγή για μια απόφαση ανταλλαγής πληροφοριών, όπου δεν πιστεύω βέβαια ότι κανείς μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι παρέχονται όλα τα εχέγγυα νομιμότητας από το σύστημα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα που έχουμε τη συμφωνία. Ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι κάθε συμφωνία ταιριάζει σε κάθε κατάσταση, αλλά στη στιγμή της την εποχή της παγκοσμιωμένης ε, οικονομίας ε, και τα φαινόμενα που έχουμε, όπως ε, αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα, ή των μεγάλων καρτέλ ή των πολυεθνικών συγχωνεύσεων, είναι ασφαλώς απαραίτητο να προωθήσουμε περισσότερες τέτοιου τύπου συμφωνίες που μπορούμε να ανταλλάσσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες. Ξέρετε ότι ήδη ε, διαπραγματευόμαστε με τον Καναδά μια αντίστοιχη συμφωνία δεύτερης γενεάς συνεχώς ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ζήτημα στη συμφωνία με τον Καναδά που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όταν απεμπλακεί το σχετικό θέμα θα σας ενημερώσουμε. Αυτή τη στιγμή ε, για άλλη συμφωνία δεύτερης γενεάς δεν έχουμε προβλέψει να διαπραγματευτούμε με άλλες αρχές, με άλλα κράτη. Πάντω είναι απαραίτητο πριν ε, να προχωρήσουμε στι διαπραγματεύσει αυτέ να έχουμε εξασφαλίσει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και σύμπτωση υποθέσεων που παρακολουθούμε ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε εχέγγυα πως ε, το νομικό σύστημα των λόγω αρχών του κράτου, προσφέρει ισοδύναμη προστασία προσωπικών δεδομένων, επίπεδο ε, ενδίκων μέσων, με αυτό το οποίο προσφέρουν και οι προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο όταν θα έχουμε ε, εξασφαλίσει πως ισχύουν όλα αυτά τα εχέγγυα θα μπορούμε να προχωρήσουμε στη πραγματεύση μιας της συμφωνίας. Το μελετούμε πάντως, ε, είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε δυνατότητες για αντίστοιχε ε, συμφωνίες δεύτερης γενεάς με άλλες αρχές, με άλλα κράτη και σταματάω εδώ για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής θέλει να λάβει και πάλι το λόγο. Ναι, να ευχαριστήσω απλώ τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πολύ καλές πληροφορίες και όπως σας είπα ελπίζω και πιστεύω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ε, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ρίσουμε το χρονοδιάγραμμα και να δούμε τον Ιανουάριο ποια θα είναι η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Ωραία. Μόλις ακούσαμε λοιπόν την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 20 ε, ε, Δεκεμβρίου, θα τις εξετάσουμε στις 9 Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 20 Ιανουαρίου και κατόπιν θα περάσει από τη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου το ζήτημα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε περίπου ένα τέταρτο στην διάθεσή μας και προσπαθούμε να βρούμε ε, τον εισηγητή για το επόμενο σημείο στην της διάταξη που είναι ο κανονισμός του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια. Καλό θα ήταν να ε, μην χρειαστεί να περιμένουμε, αλλά δυστυχώς πρέπει. Ε, πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι όταν λέμε ενδεικτικό πρόγραμμα ημερήσια διάταξη είναι όντω ενδεικτικό. Να δούμε λοιπόν αν θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ αρκετού ανθρώπου για το θέμα αυτό. Να κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα.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 Um, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καταφέραμε να τους φέρουμε όλους. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Και έχουμε λίγο επιπλέον χρόνο στη διάθεσή μας για να περάσουμε απευθείας στο σημείο 5 της ημερίας διάταξης και την πρόταση για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματογοράς. Να δώσω απευθείας το λόγο στον συγητή, τον Σαΐντ Ελκαντράουι. Σαΐντ. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου σε γενικές γραμμές, θα ήθελα να σας παρουσιάσω λίγο το πλαίσιο. επί του οποίου ε, λειτουργεί το σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μπορεί να διαβάσετε την έκθεση του Financial Stability Board ε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, από την οποία έκθεση προκύπτει ότι από το 2012 ο σκιώδης τραπεζικός τομέας αυξήθηκε κι άλλο και φτάνει πλέον στο 1-3 ε, δολάρια. 170% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος ε, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει αυτό το ποσό. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσω των όσων μας λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο τραπεζικός τομέας αυτές οι μη χρηματοπιστωτικές ε, δραστηριότητες είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστούν τα τελευταία χρόνια και πρέπει να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να περιορίσουμε τους κινδύνους ε, στο συγκεκριμένο τομέα. Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο για τα αμοιβαία κεφάλαια εμπίπτει ακριβώς αυτό το πλαίσιο, να λάβουμε υπόψη δηλαδή το σκιώδη τραπεζικό τομέα. Σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε, σας είχα πει ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μια καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις δεδομένου ότι έχουμε κάνει και εμείς κάποιες διαπιστώσεις ε, όταν εγκρίναμε τη σχετική έκθεση για τον σκιώδη τραπεζικό τομέα και προέκυψαν και μια σειρά συστάσεων από τη συγκεκριμένη έκθεση. Στο μέτρο του δυνατού προσπάθησα να λάβω υπόψη αυτές τις συστάσεις. Όσον αφορά τώρα τη δική μου την έκθεση, τα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη χρηματοδότηση των τραπεζών ε, και των δραστηριοτήτων ε, των αρχών των κρατών μελών βραχυπρόθεσμα. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να πάψει να υπάρχει αυτό το μέσο, αλλά θα θέλαμε να είναι πιο σταθερό και πιο διάφανο το όλο σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε να γίνεται μία ε, διάκριση μεταξύ των περιβόητων ΣΥΝΑΦ, των οποίων η αξία αντικατοπτρίζεται σε ευρώ ή σε δολάρια και όπου είναι ε, κειμενόμενες οι μεταβλητές ε, και ε, τα λεγόμενα ΒΙΝΑΒ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σταθερά κεφάλαια, επειδή υπάρχει θέμα διαφάνειας, τίθεται ένα ποσοστό της τάξης του 5% για το αποθεματικό και δίνονται και τρία χρόνια ε, για ένα μεταβατικό διάστημα. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι θα πρέπει να εισαχθούν αυτά τα λεγόμενα buffer που προτείνονται αμέσω, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το κεφάλαιο, το αποθεματικό του 3% μέχρι το 2014 και πρέπει αυτά τα buffers να είναι έτοιμα το συντομότερο δυνατόν. Η δική μου η πρόταση... Ε, ε, ήταν ε, μακροπρόθεσμα, ίσως σε ορίζοντα μιας πενταετίας, να πάψουμε να έχουμε ΣΥΝΑΦ και να έχουμε μόνο ΒΙΝΑΦ. Ε, αυτό δεν είναι βέβαια δική μου επινόηση. Έχει προταθεί από τους τραπεζίτες των κεντρικών τραπεζών και δεν ξέρω αν ακούσατε και τον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος στη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Επιτροπής μας ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη τάση. Ε, και στην έκθεση που είχαμε το 2012 ζητήθηκε το ίδιο και το ίδιο ζήτησε στην τελευταία της έκθεση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας των Χρηματιστήριων. Ε, η έκθεσή μου λοιπόν αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Θα υπάρξει μια μετάβαση μέχρι το 2014 και θεωρούμε ότι το πλεονέκτημα θα είναι να έχει λίγο χρόνο ο τομέας να οργανώσει όλες αυτές τις δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις να έχουν το κατάλληλο χρόνο στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν πιο ασφαλή τρόπο χρηματοδότησης. Όσον αφορά τώρα τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, το οποίο αναλύεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ και εγώ ότι είναι σημαντικό, διότι έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ε, ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που ενέχονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια. Έγινε η σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας σε θέματα οίκων ε, ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει και μια κάποια ανεξαρτησία. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο λογικό. Για μια σειρά από διαδραστηριότητε, βέβαια θα μπορούσε να έχει νόημα να χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα ε, στοιχεία και να υπάρχει και η βαθμολόγηση και το σχετικό rating από έναν οίκο πιστοληπτικής αξιολόγηση και ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι μία εκ των παραμέτρων που πρέπει να λαφθούν υπόψη. Καταλαβαίνω λοιπόν ποιο είναι το σκεπτικό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το θέμα είναι ότι το ίδιο το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να καθορίσει μία σειρά από δραστηριότητες που θα το επιτρέπει να κάνουν μία ανεξάρτητη αξιολόγηση και να κρίνουν κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί μια διαδικασία ή όχι. Ε, αντιλαμβάνομαι την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζω ε, σε κάποιο βαθμό τα όσα λέει, αλλά ίσως υπερβαίνουμε λίγο τα εσκαμμένα όταν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες βαθμολογίες που θα γίνονται για κάθε μία ε, ε, ΚΑΕ. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σειρά από σαφείς οδηγίες και η κάθε μία να αποτελεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο και από εκεί και πέρα να δίνεται συγκεκριμένη έγκριση ε, και αδειοδότηση. Έτσι θα έχουμε κάτι πιο ασφαλές. Τι άλλο πρέπει να προτείνουμε τώρα. Ίσως σε πολύ αυστηρές συνθήκες θα μπορούσαμε να ενδύσουμε σε συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια ε, και θα μπορούσε ίσως να είναι μια λύση αυτή. Τα αμοιβαία κεφάλαια βέβαια για κάποιες επιχειρήσεις αποτελούν ένα μέσο το οποίο τους επιτρέπει να κάνει μια καλύτερη κατανομή κινδύνου. Αντί να επενδύσουν σε ένα και μόνο ταμείο, ε, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να επενδύσουν σε περισσότερα. Ένα ακόμα θέμα Είτε θα έχουμε λοιπόν ε, ε, usage, είτε θα έχουμε εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Και εάν ε, εγκριθεί τη σχετική έκθεση, θα έχουμε ένα ακόμα μέσο στη διάθεσή μας. Σε περίπτωση βέλτιση βέλτιστης χρήσης, τα αμοιβαία κεφάλαια και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται φυσικά αυτά τα κεφάλαια, αν εδρεύουν σε μια τρίτη χώρα, θα πρέπει να φροντίσουν να μην βρίσκονται σε κάποιο φορολογικό παράδεισο. Όπως είχαμε ήδη προβλέψει και ε, σε αντίστοιχη νομοθεσία για τα θέματα αυτά και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλη διαφάνεια για τους μισθούς που λαμβάνουν ε, οι επικεφαλείς αυτών των ταμείων και νομίζω ότι η έκθεση του συναδέλφου για τα θέματα αυτά είναι πολύ καλή πηγή έμπνευση. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υποπτεύσουμε πολύ καλά την εφαρμογή τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν ακόμα βελτιώσει στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ευρωεπιτροπή. Και όσον αφορά τα μεγαλύτερα ε, κεφάλαια, τα οποία ε, διαχειρίζονται μέχρι και 10 δις ευρώ σε κάποιε περιπτώσει, θα πρέπει ίσω να δούμε αν θα πρέπει να γίνεται εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές λοιπόν είναι οι γενικές γραμμές ε, του σχεδίου έκθεσης μου κυρία Πρόεδρε. Ε, προσβλέπω φυσικά σε διάλογο με τους συναδέλφους και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε ένα μήνα στη διάθεσή μας για ανταλλαγή απόψεων και ε, να ψηφίσουμε την έκθεση το Φεβρουάριο. Και στη συνέχεια θα έχουμε περίπου ένα δίμηνο στη διάθεσή μας για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Η Ελληνική Προεδρία ανακοίνωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί ε, επισταμένα με το θέμα αυτό και να προσπαθήσει να το ολοκληρώσει. Για να δούμε λοιπόν αν θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε και εμείς πριν από το τέλος της θητείας μας, αλλά αυτό ακόμα είναι αβέβαιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκουζές, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ως ηθιστέ αλλά και με μεγάλη ειλικρίνεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προπαρασκευαστική του δουλειά και τις διάφορες επιλογές που μας προτείνει. Να αναλογιστούμε. Ιδιαίτερα ε, τα, οι δύο αυτοί οι τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς με διαφορετικές ε, δηλαδή σταθερές αξίες είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πιο ριζική προσέγγιση, δηλαδή προτείνει την σταδιακή κατάργηση των ε, αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερή αξίας και παραπέμπει στους οργανισμούς οποίους αναφέρεται και ο εισηγητή. Εγώ δεν παραγνωρίζω την ε, δυσκολία, τις δυσκολίες που έχει αυτή η επιλογή, δεδομένου ότι 50% ε, κεφαλαίων του ενός ε, τύπου όσο και 50% των κεφαλαίων του άλλου τύπου συναντώνται στην αγορά. Παραμένουν όμως κίνδυνοι κίνδυνοι που ενέχονται στα τα ε, αμοιβαία κεφάλαια σταθερής αξίας. Η θέση λοιπόν του συγκητή είναι λογική και πρέπει να την ε, κοιτάξουμε με προσοχή. Κατά τα άλλα, ένα θεμελιώδες θέμα είναι το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των αμοιβαίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Και εν προκειμένου θα ήθελα να επενθυμίσω πως θα ήταν ε, αντιφατικό και παράδοξο το να ζητήσουμε από την Επιτροπή μια σειρά από κανόνες που θα ισχύουν ε, για τα ταμεία σταθερής αξία, που προβλέπονται μάλλον ε, για τα κεφάλαια σταθερής αξίας και θα εφαρμόζονται και σε αυτά των κειμενόμενων αξιών. Επίσης ως προς την τιτλοποίηση. Ξέρω ότι ορισμένοι μετά την δυσάρεστη εμπειρία των ε, subprime προχωρούν με πολύ μεγάλη προσοχή στον δρόμο αυτόν. Πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα να τη τιτλοποίηση. Το γεγονός, όμως, ότι δεν έγινε σωστά η τιτλοποίηση στι ΗΠΑ γιατί στην Ευρώπη για τις πραγματικές εκλοποιήσεις, ευρωπαϊκές εκλοποιήσεις, δυσκολίες είχαμε ελάχιστες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να μην ε, ε, προχωρήσουμε χωρίς αυτό σημαντικό μέσο για την αναχρηματοδότηση της οικονομίας. Για, τις, ε, για την αξιολόγηση, το rating, πάλι θα ήταν παράλογο μετά από τρεις διαδοχικούς κανονισμούς για τις για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ε, που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους να απαγορέψουμε την ε, αξιολόγηση πλευρά τους και να εκτεθούμε σε οποιονδήποτε ανώνυμο ουσιαστικά αξιολογητή ο οποίος θα έβαζε ε, αστεράκια ή οποιοδήποτε άλλο σημάδι δίπλα στις, στα κεφάλαια αυθαίρετα. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω και να πω ότι πρέπει και να διευρυνθεί το πεδίο των επιλέξιμων κεφαλαίων και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της διαφοροποίησης ώστε τα μηδέα αυτά κεφάλαια να έχουν και την ασφάλεια αλλά και την αποτελεσματικότητα που τους αξίζει. Πάντως πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα και να ολοκληρώσουμε πριν από το πέρας της θείας μας. Ο Wolf Klintz ζήτησε συγγνώμη, αλλά θα τον αντικαταστήσει κάποιος εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το θέμα αυτό. Προσωπώ και τον Κλίντ αλλά και τον Σμιτ. Φαίνεται τη Δευτέρα είναι δύσκολο να έρθει κανείς στα Βρυξέλλας. Ο Κλίντ ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να προσέλθει αυτό προσώπος. Θεωρεί ότι ο κύριος στόχος των νέων κανόνων είναι να στα υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα. Να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τα εξής μέσα. Πρώτον, κατώτατα όρια των ρευστότητας που να πρέπει να γίνονται σεβαστά και το πολιτή πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και στη βάση των επενδυτών. Κατά τις σκιώδεις τραπεζικές συζητήσεις ζήτησε ήδη ο κ. Κλίντς από την Κομισιόν να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα. Δεύτερον, ενίσχυση της ποιότητας των πόρων. Τρίτον, να υπάρχουν τέλη ρευστότητος εάν διαπιστωθεί ασυνήθιστα υψηλός ρυθμός εξυγιάνσεων που χρειάζονται για να μπορεί το Ταμείο έτσι προσωρινά να τις πάβει. Αυτά τα μέτρα δεν διαφέρουν και πολύ από το ΆΙΟΣΟΚ. για να μπορεί το Πολδίπ να αντιμετωπίσει τις απαραίτητες εξηγιάνσεις. Και γι' αυτό ο κύριος Κλίντς σε ελαφριά διαφωνία με τον εισηγητή δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή σύγκληση για όλα. Δέχεται την πρόταση του εισηγητή να υπάρχουν αυστηρότεροι όροι γιατί η μηχανική εξάρτησή μας από εξωτερικές αξιολογήσεις και αξιολογικές εταιρείες πρέπει να μειωθεί. Πρέπει να δημιουργήσει το πολυπτικού του μηχανισμούς για την αξιολόγηση των κινδύνων και να χρησιμοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση μόνο σε τελευταίο λόγο. Επίσης πρέπει να καθορίσει ορισμένες διαδικασίες για καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επενδυτών και ιδιαίτερα της ανάγκης τους για ρευστό. Οι κανόνες διαφοροποίησης είναι σημαντικό εργαλείο για να αποφευχθεί η συγκέντρωση των κινδύνων και συμφωνεί ο κ. Κλίντς με τον εισηγητή ότι κάθε δημόσια αρχή μπορεί να πρέπει να την χάνει τέτοια στήριξης και προσβλέπει στην συνέχιση της επικοδομητικής συνεργασίας με τους Σκιώδης και με τον εισηγητή. Και το άλλο βέβαια θα ήταν ενδιαφέρον να τα πω και στα γερμανικά. Να, αλλά δυστυχώς τα έχουν γράψει στα αγγλικά και γι' αυτό σας τα διάβασα στα αγγλικά. Thank, you very much. Uh, now for the Greens, Philippe για τους πράσινους τώρα ο κύριος Λάμπερτ. Εγώ θα εκπροσωπήσω τον εαυτό μου. Ίσως να είμαι και διχασμένη προσωπικότης, αλλά δεν νομίζω. Θα παραμείνω συνεπής με τον εαυτό μου. Διχασμένη, ποιο τμήμα σας προτιμ, μου προτιμάτε. Α, μετά άλλη φορά θα το πούμε αυτό λοιπόν. Εδώ φαίνεται ότι δημιουργείται μια μεγάλη ευρεία συνένεση. Γιατί φαίνεται ότι όλοι συμφωνούν με τον Σαΐντ. Και εμείς συμφωνούμε με τις γενικές κατευθύνσεις του εισηγητού για την ιδέα ενός προοδευτικού facing out. Επίσης, για το θέμα των φορολογικών παραδείσων και τις όσο δυνατόν λιγότερης προσφυγής σε, στα ΟΤΕΣΕ. Εγώ τώρα θα περιοριστώ στα θέματα όπου θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς, διότι εάν πούμε ότι τα νομισματικά ταμεία σε σταθερές τιμές πρέπει να καταργηθούν, Ήδη καταπίπτουν πολλές από τις τροπολογίες μας. Θεωρούμε ότι τα ταμεία σε σταθερές τιμές λειτουργούν σχεδόν ως τράπεζες και άρα ότι θα πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις με τις τράπεζες. Αλλά αφού μιλάμε, αν μιλάμε για phase out, τότε πρέπει να δούμε με τι ταχύτητα θα γίνει το phase out. Και τι όριους θα επιβάλλουμε κατά την περίοδο του phase out. Όλα εξαρτώνται από τη μεταβατική περίοδο. Αν είναι σύντομη, τότε δεν χρειάζεται να βάλουμε πρόσθετους όρους. Αν όμως είναι μακρύτερη, τότε πρέπει να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για να αποφευχθούν πρόσθετοι κίνδυνοι. Επίσης θεωρούμε ότι για τα θέματα των αμοιβών πρέπει να γίνει κάποια περισσότερη συζήτηση. Για τα σχέδια recovery δεν έχουμε πει αρκετά. Πώς θα διασφαλίσουμε δηλαδή την διάσωση των ταμείων αυτών σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν ατομικά ή συστημικά προβλήματα. Συμφωνώ με τον Ζαν Πολ και για τις εταιρείε πιστοληπτικής αξιολόγησης, αλλά Υπάρχει και το θέμα των πληροφοριών που διαθέτουν ή δεν διαθέτουν τα ταμεία αυτά, άρα υπάρχει εδώ ένας ρόλος για την ΕΣΜΑ. Ανάλογο με αυτό που κάνει ανάλογη αμερικανική εταιρεία FCC, ε, υπηρεσία. Τώρα για τη ρευστότητα, όπως είπε και ο Ζαμπόλ, πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό μεταξύ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτά ήθελα να θίξω και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σύντομα πάνω στο κείμενο αυτό για να έχουμε επιτέλους τελειώσει και να δούμε επιτέλους για το shadow banking πριν λήξει η θητεία αυτή. Τώρα έχουμε ένα τέταρτο κόμμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν ε, ενημερώθηκες, αλλά είναι η σειρά σου τώρα. Πάνω στην ώρα λοιπόν ήρθα και καθυστέρησα το ακαδημαϊκό τέταρτο, τέλος πάντων ζητώ συγγνώμη. Και ζητώ συγγνώμη αν κάποια από αυτά τα οποία θα αναφέρω έχουν ήδη αναφερθεί ή κάποιο τα έχει απορρίψει ήδη οτιδήποτε άλλο. Απλά είναι αυτά τα οποία θέλω να θίξω. Μας αρέσει το γεγονός ότι ο εισηγητής ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αμοιβαία κεφάλαια ώστε να υπάρχουν δυνατότητα διαφοροποίησης σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται ε, με τα κειμενόμενα κεφάλαια δεν συμφωνούμε απολύτω με τη διαγραφή των ε, οίκων ε, αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα και δεν συμφωνούμε απολύτω ότι τα κειμενόμενα είναι πιο ευάλωτα από τα σταθερά κεφάλαια. Ε, υπάρχουν κάποια παραδείγματα για ε, ε, ε κειμενόμενα τα οποία είναι εξίσου επικίνδυνα με τα σταθερά ή το αντίστροφο. Και επίση δεν είναι μόνο 3% το αποθεματικό. Ορισμένε φορέ θα πρέπει να γίνει μετατροπή όπως προτείνεται σε 5 χρόνια. Εγώ με ανησυχεί αυτή η πρόταση. η περιορισμένη χρήση των ταμείων αυτών για βραχυπρόθεσμα ε, ε, διάστημα 90 ημερών, πολλέ φορέ και σε κειμενόμενα κεφάλαια έχουμε αντίστοιχου όρου. Εμεί είμαστε υπέρ αυστηρότερων όρων που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ε, έλλειψη κινδύνου στον ε, τομέα αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει για τεστ ε, να υπάρχουν ε, κανόνε διαφάνεια πολύ συγκεκριμένοι. Χαίρομαι επίσης που ο εισηγητή αναφέρεται σε εξωτερικούς ε, αξιολόγηση πιστολεπτικής ικανότητα, αλλά θεωρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει τα όρια όταν υποστηρίζει και το 3% του αποθεματικού και κυρίως με την απαγόρευση των ε, κεφαλαίων ε, στα σταθερής αξίας σε πέντε χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι απλώς θα κάνουμε μετατροπή από τα μεν στα δε, ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο τα χειριζόμαστε. Ε, όσοι ασχολούνται με διάφορους ε, λογαριασμούς και έχουν διάφορα κεφαλαίων να αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται και σε τι αναφέρομαι. Το θέμα είναι πού πάνε όλα αυτά τα κεφάλαια και αν θα υπάρξει εισρωή κεφαλαίων από τα ΣΥΝΑΦ, από τα σταθερά κεφάλαια στα κειμενόμενα. Αυτό που θα θέλαμε πραγματικά να υπάρξει είναι διαφοροποίηση, όχι συγκέντρωση του, του κινδύνου σε ένα κεφάλαιο και μόνον. Και νομίζω ότι έτσι θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ε, κίνδυνο μέσω διαφοροποίησης και όχι μετατροπής από το ένα στο άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος από το Ιγκού εδώ. Δεν βλέπω κάποιον εδώ στην αίθουσα. Η κυρία Λούλινγκ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από τον εισηγητή, γιατί ήρθα λίγο καθυστερημένη και δεν άκουσα τα πάντα. Δεν άκουσα ούτε καν αυτόν ούτε κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και για τους επενδυτές ε, και τους ε, θεσμικούς επενδυτές αλλά και για τους λιανικούς επενδυτές καταρχάς θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πώς έχει η κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα από πλευράς νομοθεσίας. Υπάρχουν επιτόκια τα οποία ε, φτάνουν σχεδόν στο μηδέν και τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Και γιατί αυτό. Διότι τα έσοδα και το περιθώριο ευελιξίας των ε, διαφόρων παραγόντων είναι τόσο περιορισμένα που οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή έχει συνέπειες οι οποίες είναι πολύ μεγάλου βαθμού. Τα αμοιβαία κεφάλαια πλήττονται αυτή τη στιγμή. Ε, τα επιτόκια ήταν στο 5 με 6%. Ε, η διαφορά ε, του ενός τετάρτου ή του ενός δεκάτου θα ήταν αξιοσημείωτη. Αλλά όταν είμαστε στο 0,25% ή στο 050 ε, οι αλλαγές είναι πολύ ασήμαντες. Και επίσης, καταλαβαίνω ένα αλλά είναι δυνατόν ο Ευρωπαίος νομοθέτης να θέλει να αμφισβητήσει ε, τα μέσα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρώ ότι είναι ε, πρόθεση καθενός, κανενός βέβαια αυτό. Καταλαβαίνω ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας ορισμένες φορές ε, έχει την τάση να φωνάζει εκ των προτέρων, αλλά πραγματικά θα ήθελα να επισημάνω ότι το πλαίσιο αυτό που έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και μάλιστα θα διαρκέσει και για αρκετό μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι εάν επιβαρύνουμε πολύ τους επενδυτές, οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ αρνητικές. Μια δεύτερη παρατήρηση τώρα. αφορά τα σταθερά κεφάλαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν οι κανόνες και μάλιστα ουσιαστικά. Ο κλάδος στο σύνολό του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και μάλιστα ιδιαίτερα έντονα. Όλα αυτά μας θέτουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κρίνουμε με αντικειμενικό τρόπο τον υποτιθέμενο κίνδυνο αυτών των ε, αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερής αξίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια μορφή εγγύησης της τάξης του 3% και ο κλάδος απαντά και λέει ότι θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει ε, μια μορφή έκτακτου φόρου σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι συνθήκες. Εγώ πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι η δημιουργία αυτού του τελευταίου μηχανισμού δεν θα αρέσει καθόλου στους ε, ε, επενδυτές. Και αντιλαμβάνομαι και πάρα πολύ καλή για, αυτό, για ποιο λόγο. Γι' αυτό λοιπόν και ρωτάω και γιατί επιλέγουμε αυτή την οδό και δεν ε, ε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτά τα κεφάλαια σταθερής αξίας για τους θεσμικούς πελάτες οι οποίοι έχουν αποκομίσουν οφείλη ενός τέτοιου μέσου το οποίο δεν επιφέρει πολύ σοβαρούς κινδύνους, ενώ οι ελληνικοί επενδυτές θα μπορούν να επενδύσουν σε κεφάλαια κειμενόμενης αξίας και πραγματικά εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εισηγητή, οι σκιώδεις εισηγητέ να μου απαντήσουν. Δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε ένα τμήμα του προβλήματος κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτές λοιπόν ήταν οι παρατηρήσεις μου και η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να εκφράσω τι ανησυχίε μου, χωρί να έχω ακούσει ολόκληρη την ε, παρουσίαση, γιατί έρχομαι από το αεροδρόμιο απευθεία. Ε, θέλω να πω ότι με ανησυχούν οι διατάξεις ε, για τα κεφάλαια όπως τις έχει περιλάβει στην πρόταση της Επιτροπή και στο σχέδιο όμως του εισηγητή της βλέπω. Εκατό δισεκατομμύρια ευρώ σε τέτοιου είδους κεφάλαια, μια πολύ σημαντική πηγή ρευστότητας για τις τράπεζες και το μετραπεζικό τομέα και αν επιβληθούν σε αυτά ε, εγγύησεις κεφαλαιοχικές στην Ευρώπη χωρίς αντίστοιχη ε, απέτηση και στις ΗΠΑ τότε τα αμοιβαία κεφάλαια αυτά μπορεί να αποφασίσουν να αλλάξουν έδρα. Θα ήθελα επίσης και νομίζω το Σαϊάτ το επεσήμανε, το την ώρα που έφτανα, ότι βρισκόμαστε και το λέει και στη σύστασή του ενώπιον του 2 2012 κάθετος 1 για τα αμοιβαία κεφάλαια ενώπιον μιας διατάξεως που μιλάει για την πιθανή εκροή αμοιβαίων κεφαλαίων από την Ευρώπη προς άλλα κράτη ή εναλλακτικά προϊόντα. Συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος θα είχαν βαρύτατο αντίκτυπο και στην ε, ρευστότητα και στη βραχυπρόθεσμη δυνατότητα δανεισμού για τους Ευρωπαίους ιδιαίτερα Τράπεζα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν εξετάζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να μελετήσουμε τα όσα λέει το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, μια γενική απαγόρευση θα είχε συνέπειση όχι μόνο προ την απασχόληση αλλά και το εθνικό εισόδημα, αλλά και απώλεια ρευστότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών που δεν, μπορούμε, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι είδους ε, συνέπειες θα φέρουν. Και έτσι παρακαλώ την Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς των Πολιτειών για εναλλακτικέ με ε, τέλη ρευστότητα και ασφαλιστικέ δικλείδε, που είναι πιο λογική και πρακτική για μένα. Είναι μια λύση δηλαδή που επιτρέπει και ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ενώ, οντοτήτων, ΗΠΑ και ΕΕ και πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά. Συμφωνώ με τους άλλους συναδέλφους που επισημαίνουν την ιδιαίτερη αυτή δυσκολία και πιστεύω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να μελετήσουμε, να εξετάσουμε και αυτή τη λύση. Για να μην πούμε σαν τάβρος ή άλλο πολύ όπως λέμε, πρέπει προσεκτικά να μελετήσουμε τις συνέπειες της όποιας επιλογής μας, γιατί υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Θέλω και εγώ να τοποθετηθώ, λέει η Πρόεδρος. Και σας καλώ να κοιτάξετε στην ε, ιστοσελίδα της ε, Επιτροπής μας ομιλίες μου στη διάσκεψη γιου τη πρώτη που έχει να κάνει με τα κεφάλαια και μια άλλη ομιλία στην ε, διάσκεψη που αφορά την διασφάλιση και την ε, τίτλοποίηση που ανέφερε ο Ζων Πολ. Εγώ νομίζω ότι προτιμώ τα αμοιβαία κεφάλαια και όχι την τίτλοποίηση τόσο πολύ. Τη σωσιακά καλύτερα μάλλον, αντί για τη τίτλοποίηση. Ε, ας τα κοιτάξουμε λοιπόν και ας κοιτάξουμε πολύ προσοχή τι είδους, ε, σε, σε πόσα κομμάτια θα κόψουμε αυτά τα κεφάλαια. Η εναλλακτική στη ΣΟΣΕΚΑ δεν είναι σαφέ ε, τι μορφή θα πάρει σε διάφορε κράτηπε, εάν τα χρήματα πάνε σε, άλλα κράτη, αν τα χρήματα πάνε σε τράπεζε, καθώ είμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από αυτέ, ίσω δεν είναι τόσο κακό. Ή μπορεί να μετατραπούν σε λιγότερο ρυθμισμένα προϊόντα. Άρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι του γάτα με το ποντίκι. Ή μπορεί να εγκαταλείψουν την έδρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο διόλου. Ιδιαίτερα κάποιοι επενδυτέ μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, τράπεζες, χορηγοί που συνηθίζουν να σηκώνουν το χρήμα τους και να το μετακινούν πάρα πολύ γρήγορα. Άρα δεν πρέπει να μόνο ότι υπάρχουν και άλλου τύπου άξιοι επενδυτές για στέγη, για κοινωνική στέγη, για υποστήριξη κοινοφελούς έργου κτλ. που ίσως να μην μετακινηθούν τόσο γρήγορα. Αυτοί είναι που θα υποφέρουν περισσότερο, θα αναγκαστούν, θα πιεστούν προς πιο ε, ρηψοκίνδυνα προϊόντα, ενώ οι, οι, οι, πιο σκληροί επενδυτές δεν θα, θα διστάσουν να φύγουν γρήγορα. Αυτοί λοιπόν οι επενδυτές που μας μοιάζουν θα λέγαμε, που θέλουμε να υποστηρίξουμε, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Άρα και εγώ θα υποστηρίξω την πρόταση να κοιτάξουμε λύσεις, ε, δυσφαλιστικές δικλίδες, τέλη που θα λαμβάνουν υπόψη και την ρευστότητα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν κάποιοι διοικητές κεντρικών τραπεζών έχουν πει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά, αλλά αν δούμε τα ΟΣΕΚΑ ΣΥΝ με όλες τις προϋποθέσεις που συνεπιφέρουν. Ε, δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην ε, ζημιώσουμε κανέναν από αυτούς που μας ενδιαφέρουν. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου άσπρο μαύρο αυτή η υπόθεση και έχω ήδη πει ότι ναι, είναι παράξενο στην Ευρώπη να λέμε ότι θέλουμε την τυπλοποίηση αφενός αφετέρου, δεν την απαγόρευση των ΟΣΕΚΑ. Και δεν υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να ελέγξουμε και τις δύο επιλογές και γι' αυτό παρακαλώ τον εισηγητή πολύ προσεκτικά να σκεφτεί, να ξανασκεφτεί τους περιορισμούς και την ιδέα για απαχώρευση που προτείνει. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή λύση. Πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε και πρέπει να πω ότι ομιλώ χωρί διαβούλευση με την ομάδα μου. Αλλά, εν πάση δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να περιχαρακωθούμε σε κομματικές γραμμές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε για τον Ευρωπαίο επενδυτή, εκείνον το μικρό επενδυτή που έχει παγιδευτεί, που δεν μπορεί να στραφεί πουθενά αλλού και δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, καταστρέψουμε ευκαιρίες, καλές επιχειρησιακές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να ε, κάνουμε κακό στις δικές μας επιλογές χωρίς να έχουμε βρει μια λύση ασφαλή και αποδοτική προηγουμένως. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει το λόγο. Ας την ακούσουμε και μετά ακούμε τον Σίγητα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα και μια σύντομη έγκριση θα ήταν το καλύτερο για να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να αναλάβει τις ευθύνες της για αυτό το θέμα του shadow banking. Η έκθεση του εισηγητή είναι επίκαιρη και προκύπτει από μακρές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, πράγμα για το οποίο τον συγχαίρουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Στην πρότασή μας ζητούμε αυστηρούς κανόνες, γιατί είδαμε κατά την κρίση ότι δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν τα ταμεία της πιέσεις των αγορών και οι κανόνες αυτές 5 με 10% διαφοροποίησης και ορισμένο κατώτατο όριο ρευστότητας είναι στοιχειώδης. Τώρα, για τις εταιρείε αξιολόγησης πράγματι ο κανονισμός που ισχύει έχει βελτιώσει πολύ τα πράγματα και την ποιότητα των βαθμών που έβαζαν, αλλά Κατά τη δική μας αξιολόγηση διαπιστώσαμε ότι τα ταμεία με σταθερές αξίες, τα ΣΕΝΑΒ που λέμε στη Γαλλία, είχαν πρόβλημα. Μόνο το τριπλό α προβλεπόταν ως βαθμολόγηση και τίποτε άλλο. Άρα δεν... αυτό προκύπτει από το ότι είναι σχεδόν εγγυημένα αυτά τα ταμεία, αλλά μόλις καταργήθηκε αυτή η βαθμολόγηση, σημειώθηκε μεγάλος πανικός. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι η καλύτερη λύση ήταν να καταργηθεί αυτή η βαθμολόγηση γιατί τα ταμεία αυτά ούτως ή άλλως λειτουργούσαν άψογα. Τώρα για τα τέλη σε περίπτωση που δεν, υπάρχουν δεν υπάρχει εγγυημένη ρευστότητα κάνουμε αυτό που κάνει και η SEC στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά διαπιστώσαμε ότι τέτοια μέτρα υπήρχαν ήδη και στην Ευρώπη γιατί ήδη είχαμε το δικαίωμα να καταργήσουμε χρηματοδότηση, να σταματήσουμε χρηματοδότηση ή να επιβάλλουμε κυρώσεις και έχει χρησιμοποιηθεί από τα Ταμεία σταθερής, ε, Σταθερών Αξιών. Γι' αυτό και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, το έβαλαν στην επίσημη νομοθεσία τους. Εμείς δεν χρειάζεται νομίζω αφού υπάρχει ήδη. Τώρα για το ερώτημα ως προς τους θεσμικούς επενδυτές και τους ιδιώτες επενδυτές υπενθυμίζουμε απλώς τους αριθμούς. Η θεσμική είναι 95% των ε, ποσών που έχουν εναποτεθεί στα ταμεία σταθερών αξιών. Οτιδήποτε και να προβλέπαμε για τους ιδιώτες δεν θα άλλαζε η κατάσταση ως προς τους συστημικούς κινδύνους. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να βρω πολλές απαντήσεις σε αυτό, αλλά ας τα πει ο καλύτερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά περιμένω τις τροπολογίες σας όλων και είμαι πεπισμένος ότι με εκείνε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Ο μου στόχος παραμένει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Επίσης έχω την εντύπωση ότι το βασικό στοιχείο της συζήτησης είναι τα μία σταθερής ή όχι αξίας. Και ξέρετε ποια είναι η θέση μου σχετικώς, την είπα πριν. Επενθυμίζω ότι για μένα τα, τα μία αυτά, τα ποσά αυτά σταθερής αξίας πρέπει να καταργηθούν ώστε οι επενδυτές να βρουν άλλες λύσεις. Ίσως από το τραπεζικό σύστημα. Αλλά αυτό ίσως αφορά λίγους μόνο επενδυτές ή για κρατικά ομόλογα, με κρατικά ομόλογα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο φόβος που εκφράστηκε για τις επιχειρήσεις που θα έφευγαν από την Ευρώπη δεν μου φαίνεται δικαιολογημένος γιατί η νομοθεσία στοχεύει ακριβώς στο ότι θα καλύπτονται και οι διοικητές των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων όπως και οι υπόλοιποι πελάτες των ταμείων αυτών. Βέβαια δεν έχει λήξει πλήρως η συζήτηση αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μερικοί ζητάνε να καταργηθούν αυτά τα ταμεία σταθερής αξίας. που επενδύουν αποκλειστικά σχεδόν κρατικά και γι' αυτό ζητούμε να καταργηθούν. Η συζήτηση λοιπόν δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, ούτε έχουμε ξεφύγει από την πραγματικότητα και αλλού τα συζητάνε αυτά. Επίσης υπενθυμίζω ότι πολλοί διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι, έκαναν ανάλογες προτάσεις όσα και πρέπει να τις λάβουμε και εμείς υπόψη μας στην νομοθετική μας εργασία. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να δηλώσω προς τον συνάδελφο Γκοζές ότι πρέπει πράγματι να ξαναδούμε τους κανόνες για τη ρευστότητα. Έχετε δίκιο. Όταν ζητάτε καλύτερη, σωστότερη εξισορρόπηση μεταξύ ασφάλειας και πραγματικής συμφέροντος της πραγματικής οικονομίας θα επανέλθω όταν συζητήσουμε τις τροπολογίες. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε η πρώτη ανταλλαγή λοιπόν απόψεων και η εξέταση του σχεδίου είναι σήμερα 2 Δεκεμβρίου, έγινε και αυτό. Η διορία κατάσταση των προγειών λήγει στις 5 η ώρα στις 10 Δεκεμβρίου. Θα τη συζητήσουμε 20 Ιανουαρίου με στόχο να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας 12 Φεβρουαρίου, άρα στην Ολομέλεια τον Απρίλιο μάλλον. Τώρα η Κομισιόν επίσης βιάζεται, αλλά δεν είναι πιθανόν να καταφέρουμε να ο τριμερής διάλογος και να τελειώσει νωρίτερα. Εκτός αν το Συμβούλιο συμφωνήσει απολύτως και η Κομισιόν γνωρίζει ότι αφού δεν έκανε τις προτάσεις πριν το Σεπτέμβριο έτσι θα πήγαιναν τα πράγματα και εμείς έχουμε ζητήσει να μας τα υποβάλει νωρίτερα αλλά ειλικρινά εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω βαρεθεί πια να μας καθυστερούν και μετά να μας λένε ότι πρέπει να βιαστούμε. Γιατί έτσι θα γίνουν οι εξετάσεις μας πρόχειρα και χωρίς την απαραίτητη διαφάνεια. Θα εργαστούμε όσο σκληρότερα και γρηγορότερα μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να προχειρολογούμε. Εμείς ούτως ή άλλως εργαζόμαστε ταχύτερα από την Κομισιόν. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Το 6. Δεν είναι εδώ ο Hans Peter Martin. Βέβαια θα περιμένουμε ο λίγα λεπτά μέχρι να τον βρούμε τον εισηγητή και τους σκιώδεις για το επόμενο θέμα. Jean-Paul, juste poser... Jean-Paul, question, ερώτηση, κυρία Πρόεδρε η ψηφοφορία θα γίνει στις 5, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πάνε κι αλλού και θα ήθελα να ξέρω αν θα γίνει ψηφοφορία στις 5. 5. Ναι. Θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον για την ψηφοφορία. Αλλά αν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας πριν από την ψηφοφορία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την έκθεση για την ενίσχυση της συνοχής των ε, ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα μπορούσε ίσως αυτό να αφορά το Προεδρείο και τους συντονιστές. Ε, να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν λίγο το χρόνο μας και να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για αυτά.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

Jean Paul. Γνωρίζουμε κάτι για τον Αλφρέντο, γιατί δεν μπορούμε να τον βρούμε. Θα έρθει ή θα μιλήσει εσύ εκ μέρους του. Δεν ξέρει τίποτα να μα πει. Δεν γνωρίζω. Αν πρέπει όμως μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του, να πω ότι συγχαίρω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και λοιπά και λοιπά. Oh, Κυρία Πρόεδρε, από ό,τι μου λένε ο κύριος Μπέρτο θα αντικαταστήσει τον κύριο, Παλό, τον κύριο Παλώνε. Ο κύριος Μπέρτο είναι εδώ. Ο κύριος Μπερτό είναι εδώ. Θα έρθει. Θα αντικαταστήσω τον κύριο Μπερτό εγώ αν δεν έρθει. Um, πιέζουν από όλες τις πλευρές, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται, παράλληλες επιτροπές. Θα έλεγα λοιπόν να προχωρήσουμε το σημείο 6. Και αν ε, χρειαστεί να ακούσουμε τους ε, σκιώδεις χωρίς να είναι σειρά τους, ας το κάνουμε και αυτό, ή ο Ζαν θα αναλάβει τα ενία. Λοιπόν, έχουμε τι. στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών. Όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατά εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέση ορισμένων μέτρων. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Hans Peter Martin, έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ στομό στα αγγλικά. Και τι... Είναι απλό, καθώς είναι απλό το πράγμα. Ας περάσω στο γερμανικό, όμως, για να προχωρήσουμε και λίγο πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Τεχνικό θέμα περισσότερο. Για όλους αυτούς ε, που συνεργάστηκαν θα ήθελα να έχω τις ευχαριστίες μου. Ιδιαίτερα αναφερόμαστε και στην ομάδα της ε, Επιτροπής, αλλά με, τους, με τον είχαμε πολύ καλό συντονισμό, αλλά και στους κοιόδης. Έχουμε εδώ να κάνουμε με μια επιδίωξη η οποία δεν ε, ικανοποιείται 100% γιατί έχουμε αρκετά μεγάλες διαφορές ως προς την ποιότητα των στατιστικών ε, ε, δεδομένων μεταξύ αφενός με των συντηρητικών Βρετανών, αφετέρου σοσιαλιστών και δημοκρατών, φιλελευθέρων και άλλων. Προσπαθούμε να κάνουμε συμβαστικές τροπολογίες, α, διαφορετική υποδοχή και υποστήριξη είδαμε σε ένα βαθμό με ξαφνιάστηκε όμως ότι κάποιοι είπαν ότι αν δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα φορολογικών αρχών θα απόσχουμε. Και από την άλλη γίνεται μια έκκληση να αναπτύξουμε τις επαφές μας και τις διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσουμε 26 μέλη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού δεν έχουμε εδώ παρόντες. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 5. Ίσως μέχρι τις 5 κάποιοι να έρθουν. Δεν ξέρω σκιώδεις αν μπορέσουν και να λάβουν το λόγο βεβαίω. Και τέλο πάντων, διευκρίνω λίγο την κατάσταση. Πάντως, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική συνεργασία. Okay, that was... Ευχαριστώ πολύ. Όντω, πολύ γρήγορα μας τα είπατε. Ζων Πολ, θες τώρα το λόγο. Θε αργότερα. Πρόεδρε, αφού δεν έχει φτάσει και ο συνάδελφος, δεν έχω τίποτα να πω εγώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του, ως ήθιστε. Εδώ. Και βεβαίως ό,τι έχει διαπραγματευτεί ο σκιώδης για τις ε, συμβαστικέ μα τροπολογίε, αναλόγω και θα ψηφίσει η ομάδα μας. Η πρόεδρος. δεν βλέπω. Α, όχι, όχι, έχουμε ακόμα έναν ε, μια καλή και πιστή απομίμηση του Όριου Σμιτ. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να αρθώ στο ύψο των περιστάσεων. Μην το το πείτε όμως. Το σχόλιο του κυρίου Πέτερ Μαρτίν δεν ακούστηκε. Μπορεί να παρεξηγηθεί. Όλοι λοιπόν θέλει να ευχαριστήσει τον Χάνς Πέτερ Μάρτιν και τους λοιπούς και όδης εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά και τη βούληση για συνεργασία. Τον ικανοποιούν συμβαστικέ τροπολογίε. Ε, είναι ευγνώμων για το γεγονό ότι πολλέ από τι δικέ του προτάσει ενσωματώθηκαν σε αυτέ. Είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την συλλογή στατιστικών δεδομένων η έκθεση αυτή χωρί επιπλέον διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα μικρομεσαίων που μπορεί να προξενήσει επιβραδύνσεις στην οικονομία και προβλήματα. Ιδιαίτερα είναι ικανοποιημένο ο κύριο Σμιτ για το γεγονό ότι μπορούσατε να καταλήξετε συμφωνία για διάφορα ζητήματα, ιδιαίτερα την ανταλλαγή των απόρριτων πληροφοριών. Εκεί υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα. Το απόρριτο των στατιστικών, η θεμελιώδης αρχή των ευρωπαϊκών στατιστικών πρέπει να γίνεται σεβασμό, Προβλέπεται στον κανονισμό 223 για τη διαβίβαση ε, στατιστικών και απορρίτων στοιχείων, εάν δεν είναι ε, βέβαιες για την ε, προστασία του απορρίτου των στοιχείων που προσφέρουν στατιστικές υπηρεσίες ή επιχειρήσεις, αν δεν είναι βέβαιες ότι μόνο για στατιστικούς λόγους θα αξιοποιηθούν, ότι θα είναι προστατευμένες από προσβολή αυτού του απορρίτου, δεν θα συνεργάζονται καθόλου ενδεχομένω στο μέλλον και θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και τις προτάσεις της εποπτικής αρχής ε, πριν να μιλήσουμε για το πεδίο εφαρμογής και το εύρος αυτής της οδηγίας. Ε, προτείνουμε να καταψηφιστεί το σχετικό τμήμα της σχετικής τροπολογίας στο δεύτερο κομμάτι για τη χρήση για, τις ε, για στατιστικό λόγο διαφτήρηση των στοιχείων μπορεί να γίνεται κατά τρόπο εθελοντικό, αλλά μόνο για κατά μέγιστο πενταετή ε, κατα, ε, κατακράτηση των στοιχείων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Ε, όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος μπορούμε να συμφωνήσουμε στην παράταση της ανταλλαγής των απόρριτων πληροφοριών. Είναι βέβαια ο κ. Σμίτ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Σας καλεί να υπερψηφίσει την τροπολογία υπαριθμών 19 για την ε, συλλογή μόνο από τον έναν εκ των δύο εισαγωγέα ή εξαγωγέα των ε, στοιχείων των σχετικών με εξαγωγές, ε, συγκεκριμένα τον εξαγωγέα, για λόγους απλούστευσης και αποφόρτησης διοικητικής. Σας ευχαριστώ. Καλώς λέει πρώτος ευχαριστώ. Το ΕΛΚ, κύριε Πόστος. Μιλώ εξ ονόματος ε, και του κύριου Παλώνε, ο οποίος παρακολούθησε το θέμα αυτό εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ τον κύριο Μάρτιν και όλους τους σκιώδεις εισηγητές ε, για ό,τι έκαναν. Πρόκειται για μια εκθέση ιδιαίτερα τεχνική, η οποία δεν είχε προβλήματα από πολιτική σκοπιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασε τον κανονισμό που σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών υπό το φως του νέου θεσμικού πλαισίου που καθορίστηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να έχουμε πράξη κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και μια πλήρη αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στατιστικών για τα ε, κεφάλαια μέσω μιας νέας ε, δομής που θα αντικαταστήσει την ε, παρούσα Επιτροπή Ίντραστατ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή, αλλά προσπαθήσαμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Μέσω των τροπολογιών μας θέλουμε να επισημαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι πράξει κατεξουσιοδότηση να, έχουν, να μην έχουν επιπλέον διοικητικό άχθο για τα κράτη-μέλη και η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων να γίνεται με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση από οικονομική σκοπιά για τα κράτη-μέλη. Επίση, προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιε τροπολογίε για να βελτιώσουμε το κείμενο όσον αφορά τη δομή του στατιστικού συστήματο ε, για την καλύτερο ορισμό των στατιστικών αξιών και στην αξία του να έχουμε εναρμονισμένους και απλουστευμένους κανόνες για την ε, διαβίβαση δεδομένων μεταξύ κρατών μελών. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το εμπόριο αγαθών. Ευχαριστώ τους υπολείπους συναδέλφους που έχουν βελτιώσει το κείμενο με τις προτάσεις τους και η μόνη επίκριση που μπορούμε να κάνουμε αφορά την αντιλαγή των εμπιστευτικών δεδομένων που είναι κάτι το οποίο προκύπτει από αυτή την αναθεώρηση ως καινοτομία. Σε γενικές γραμμές ε, μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως, αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την ανταλλαγή αυτών των δεδομένων. Πρέπει να είναι σαφές ότι η ανταλλαγή αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται μόνο για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον έχει αποδειχθεί η ανάγκη τους. Επίσης δεν θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων και για άλλους σκοπούς, ε, είτε σχετίζονται αυτοί με την φορολογία ή απλά και για ερευνητικούς λόγους όπως έχει προταθεί. Επιπλέον θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η ανταλλαγή αυτή θα πρέπει να γίνεται με εμπιστευτικό αυστηρά τρόπο και χωρίς καμία διαρροή πληροφορών προς άλλους διεθνείς οργανισμούς ή προ ερευνητικά κέντρα. Πέραν αυτού του σημείου, συμφωνώ με τι συμβιβαστικές προτάσει τι οποίε έχουμε καταλήξει με του υπόλοιπου συναδέλφου και θεωρώ ευπρόσδεκτη την πρόταση του κυρίου Σμιτ να περιορίσουμε την ανταλλαγή απόψεων χρονικά και να είναι θελοντική αυτή η ανταλλαγή. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, for the... Ευχαριστώ πολύ ο Σαΐντ για το ECR για την Ευρώπη των Συντηρητικών Δημοκρατών. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα είμαι και εγώ λακωνικός, ε, διότι δέχτηκε τις περισσότερες τροπολογίες που προτείναμε. Ε, κυρίως αυτές που υποβάλαμε με τον συνάδελφο, ένδειξη μεγάλη ενότητος ε, του κόμματος, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για ακαδηματικά ιδρύματα στις ε, πληροφορίες αυτές, σεβόμενοι ταυτόχρονα και το απόρριτο. Υπάρχουν κάποια τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, όλα αυτά δεν ε, αποτελούν πρόβλημα. Θα ήθελα να θέσω το εξή όμως. Υπάρχει μια τροπολογία για να υπάρχει ε, βεβαιότητα ότι υπάρχει συμμόρφωση με τη γενικότερη διαδικασία επιτροπολογίας, από ότι φαντάζομαι δεν θα γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία, θα έχει τους λόγους του εισηγητής. Κατά τα λοιπά σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε εδώ κάποιο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να λάβει το λόγο. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, σας παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε γενικές γραμμές καλωσορίζει το σχέδιο έκθεσης και την υποστήριξή σας ε, στην πρότασή μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η συζητήσεις που θα ακολουθήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας στο ένα ακαθόδε ζήτημα, την τροπολογία 32 και τη σχετική τροπολογία 33, που προβλέπει την ε, χρήση εμπιστευτικών ε, δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς. Αυτό δεν συνάδει με τις διατάξεις περιαπορήτου του βασικού κανονισμού για τα στατιστικά στοιχεία, των 223, και ε, με καμία γνωστή στατιστική πρακτική. Επίσης, δεν συνάδει με την τροπολογία υπαριθμών 8 του εισηγητή. Όσον αφορά κάποιες άλλες ε, τροπολογίες, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν περαιτέρω στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις και να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Κυρίως την αποδοτικότητα προς το κόστος των στατιστικών στοιχείων και αυτά θα πρέπει να εφηγραμμίζονται με τον κανονισμό 223 και με τον κώδικα δεντολογίας και καλών πρακτικών. Επίσης έχουμε το θέμα της εμπιστευτικότητας των στατιστικών στοιχείων, την τροπολογία 10 δηλαδή, και σε αυτή την περίπτωση θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή, διότι μπορεί να υπάρχουν ασυνέπειες με σχετικούς στατιστικούς κανονισμούς και να μην λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι ε, η εμπιστευτικότητα θεωρείται από τους χρήστες έως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Τρίτον, τα θέματα εκχώρησης εξουσιών, κυρίως οι τροπολογίες 14, 43, 44 και 45, επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν ακολουθείται η κοινή συνεννόηση και η θεσμική συμφωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θα εξετάσει ενδελεχώς όλες αυτές τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο συγκεκριτής θέλει να λάβει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, καταπλήσει αυτό που άκουσα από την Επιτροπή. Ε, αυτή είναι η δουλειά των, των διαπραγματεύσεων. Όταν έρθει η ώρα λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε και τα θέματα που επισημαίνεται. Καλώ λέει ο Πρόεδρος, εξετάσαμε και τις τροπολογίες. Στις 5 σε λίγη ώρα ψηφίζουμε για να είμαστε έτοιμοι για την ε, Ολομέλεια του Απριλίου. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι ώρα θα ψηφίσουμε γιατί είναι, στο, είναι καθοδόν όλοι οι συνάδελφοι. Και μια και έχουμε κερδίσει μια ώρα, προτείνω να προχωρήσουμε στη δική μου έκθεση ενίσχυση της συνοχής της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θέμα που έχει απασχολήσει μέχρι τώρα ουσιαστικά το Προεδρείο μόνο. Και αν δεν το ολοκληρώσουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και μετά την ψηφοφορία. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο να μην χάσουμε άλλο χρόνο. του υπόβαθρου. Έχει γίνει στο πρώτο ήμιση του 2013 ο δημόσιος διάλογος, η διαβούλευση για τις ε, προτάσεις ε, για την νομοθεσία αυτή. Έχουμε ετοιμάσει εμείς τις ε, ερωτήσεις, τις υποβάλαμε και λάβαμε απαντήσεις από 86 είτε άτομα είτε φορείς Δημοσιεύονται αυτές στην ιστοσελίδα, στον ιστότοπο της ε, Επιτροπής μας και προετοιμάζουμε άτυπη έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται το θέμα να φτάσει μέχρι την Ολομέλεια, αλλά διατυπώνουμε συμπεράσματα. για το σχέδιο αυτό, το οποίο θα ψηφίσουμε βέβαια, και θα αξιοποιήσουμε στο υπόλοιπο έργο μας ή σε έργο που θα αναλάβει η προσεχής ε, Επιτροπή μετά τις εκλογές. Έχω συντάξει την έκθεση με την συνδρομή της ε, γραμματείας ή καλύτερα η γραμματεία συνέταξε την έκθεση και εγώ απλώς ε, τους προσέφερα την υποστήριξή μου. Έχουμε να κάνουμε εδώ με τις απαντήσεις που δόθηκαν, ανησυχίες που εκφράστηκαν ε, και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε στα όσα επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες. Ιδιαίτερα επισημένο, επισημένονται επικαλύψεις ή αντιφάσεις στην νομοθεσία και έτσι καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετά πολύ πιο προσεκτικά την αξιολόγηση επιπτώσεων και τις, ε, και συνέπειες που μπορεί να έχει η νέα νομοθεσία που εισάγει. Ιδιαίτερα οι ενδεφερόμενοι αναφέρονται σε ανησυχίες για είτε κατακαιρματισμένα νομοθετήματα, είτε ε, αντιφατικά μεταξύ τους. Το πρίψ και το μύφιντε επί παραδείγματι. Ε, και γι' αυτό μας λένε ότι θα ήταν προτιμότερο κομμάτια της νομοθεσίας να την χάνουν επεξεργασία ταυτόχρονα. Ε, η ανάπτυξη νέας νομοθεσίας επίσης ε, θεωρείται πιο δυσκολημένα, αλλά ε, μας λένε ότι θα τους προσφέρει περισσότερη ασφάλεια. Και γι' αυτό θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει ένα δωδεκάμινο από τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας για τις τεχνικές προδιαγραφές και ταυτόχρονα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν μια, ένα σχεδιασμό προτεραιοτήτων για την νομοθεσία με αντίστοιχα κομμάτια, σχετικά δηλαδή ε, νομοθετήματα. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να ορίσει τη σειρά τέτοιου είδου νομοθετημάτων. Εμείς από πλευρά μας στο Κοινοβούλιο κάνουμε τη σχετική ε, πρόταση, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές λιγότερο. Επίσης ζητείται από τους απαντώντες συνοχή, όχι μόνο προς το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά και ως προς τους ίδιους τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς που έχουν υιοθετήσει τα μεγαλύτερα ε, κράτη. Έτσι λοιπόν ε, στο προσεχές ε, κοινοβούλιο, στην επόμενη θητεία, θα πρέπει να αποδεθούμε και σε αυτή την προσπάθεια για να δούμε και σε σχέση με τρίτες χώρες τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια άλλη ανησυχία αφορά τον, το θέμα του του συντονισμού, καλύτερου συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την Γενική Διεύθυνση για την ε, ε, αγορά, την ιστορική αγορά και μεταξύ άλλων γενικών διευθύνσεων. Θέματα που και εγώ ήδη έχω πολλέ φορέ επισημάνει, αλλά και άλλοι συνάδελφοι και που έχουν να κάνουν και με τον ε, και που έχουμε διατυπώσει και κατά τις ακροάσεις εν ώψη του, της ανάληψης των καθηκόντων των επιτρόπων. Ζητείται περισσότερη διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούνται οι συμβαστικές τροπολογίες και αρκετοί ζητούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ε, και επικοινωνίας με τους εισηγητές. Η έλλειψη χρόνου συμβάλλει πάντα στην ε, επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Τα θέματα αυτά ασφαλώς στο μέλλον θα πρέπει να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν. Για να βελτιωθεί η επισκόπηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κατάστασης και της εφαρμογής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη πρέπει να ζητούμε από τη Γενική διευθυνση Αγοράς ε, εκθέσεις τακτικές για την υλοποίηση αυτής της ε, ε, νομοθεσίας. Έχουμε βέβαια δει κάποιες ενημερώσεις σε σχέση με συγκεκριμένα νομοθετήματα που προχωρούν προς ρυθμιστική προς ρύθμιση ε, τεχνικών προδιαγραφών, αλλά θέλουμε καλύτερη ε, υλοποίηση και επαλήθευση αυτής. Επίσης, κάποιες προτάσεις αναφέρονταν σε ένα μόνο νομοθέτημα ή ένα κώδικα για την νομοθεσία, ε, πρόταση που εμπνέεται πιστεύω και από τα σχόλια ορισμένων για το ότι θα πρέπει να έχουμε έναν νόμο, ένα νομοθέτημα τύπου Dodd Frank Κάποιοι θεώρησαν ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η ιδέα, κάποιοι άλλοι βέβαια μας λένε ότι ίσως να μην είναι εφικτό ένα τέτοιο εγχείρημα και ίσως το κόστος του να είναι πολύ ψηλό. Φιλόδοξο βέβαια το έργο αυτό και εγώ προσωπικώς ανησυχώ ιδιαίτερως γιατί δεν θα ήθελα να ε, επιδεινωθεί η κατάσταση και να εισαχθεί ναι, επιπλέον παράγων αβεβαιότητας προς την νομοθεσία. Πάντως έχουμε δηλώσει ότι θα ζητήσουμε αξιολόγηση πιθανών μοντέλων συντονισμού ή κωδικοποίησης της νομοθεσίας για να έχουμε ε, μία ε, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τα γνώσεως στο θέμα αυτό. Περίμενα τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για το συνέχεια αυτών των προτάσεων και η νέα Επιτροπή μετά τις εκλογές φαντάζομαι θα βρει χρήσιμο το έργο αυτό όταν αναλάβει τα καθήκοντά της στην επόμενη θητεία. Ήταν, πιστεύω, σημαντικό το έργο που έγινε. Πολλά έχουμε να διδαχθούμε ασφαλώς για την βελτίωση του συντονισμού. Υπάρχουν αρκετές ρήτρε αναθεώρησης σε πολλά από τα νομοθετήματα και σε αυτό εντοπίζονται ορισμένε προτάσεις που μιλούν για καλύτερο συντονισμό τον αναθεωρήσεων αυτόν, Νομίζω ότι αυτό δεν είναι άσκοπο, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται. Επισήμω, ο κύριο Γκίγκολτ μόνο ενώ είναι σκιώδη ηγητή εδώ. Δεν ξέρω αν ο Ζων Πολ Γκοτζέ θέλει και αυτό να κάνει σχόλια εκ μέρου του Ελκ. Έτερο, όχι. Σβέν, έχει το λόγο. Thanks, Sharon, for, for drafting this. Ευχαριστώ, Σάρων, για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ θετικό ότι προχωρούμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το αποτέλεσμα όμως, τα συμπεράσματα ποιος και πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Παραδείγματο χάρη ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε τι φρονεί η Κομισιόν για όλα αυτά. Από τη διατύπωση Βλέπω ότι είναι πολύ θετικό που έγινε η διαβούλευση, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι τις απόψεις των ενδιαφερομένων πρέπει να τις βάλουμε στην προσθήκη στο παράρτημα του ψηφίσματος, γιατί αυτό θα αμφισβητούσε το συμπέρασμα, άμα δούμε ιδίως τη σύνθεσή τους και γι' αυτό θα το πρόσεχα πολύ. Δεν έχει ξαναγίνει εξάλλου. Ως προς την ουσία τώρα, Συμφωνώ λίγο πολύ με τις προτάσεις σου. Είναι χρήσιμες. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να δούμε μερικά πρόσθετα στοιχεία. γιατί θίξαμε το διαδικαστικό και χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια για το επίπεδο 2 και τα συμφωνώ, αλλά επίσης και για είναι σημαντική και η διαφάνεια ορισμένων τρίτων μερών όπως τους λομπιίστες. Καλό θα ήταν λοιπόν να συζητήσουμε μεταξύ μας σε περισσότερη λεπτομέρεια για να δούμε αν, αν είναι σωστό να υπάρχει τόσο λεπτομερής νομοθεσία για όλα και ποιος είναι ο ρόλος της νομοθεσίας των αγορών. Ας πούμε, αν υπάρχει ένα σύστημα μεγαλύτερης λογοδοσίας ή αποζημιώσεων, ένα σωστότερο σύστημα και αυστηρότεροι κανόνες εφαρμογής. Θα ήθελα λοιπόν ως τελικό αποτέλεσμα να γίνει μία ακρόαση ίσως με την Κομισιόν αλλά και συζήτηση μεταξύ μας γιατί οι λεπτομέρειες είναι τόσο πολύπλοκες και τόσο πολλές που μπορεί να υπάρξουν αμφισβητήσεις για μερικά. Αν δεν υπάρχει ευρεία κεφαλαϊκή βάση, ίσως θα έπρεπε να μην περιοριστούμε και εμείς σε ένα σύστημα που βασίζεται απλώς σε κίνητρα και αποζημιώσεις της αγοράς. Μια πιο ουσιαστική συζήτηση λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρουσα και σε αυτό το επίπεδο. Προσβλέπω και εγώ στο αποτέλεσμα και να δούμε τι θα το κάνουμε και πώς θα το χρησιμοποιήσει η επόμενη θητεία. Κανείς άλλος για το ίδιο δεν βλέπω. Ευχαριστώ πολύ Σβέν. Ίσως να συζητήσουμε περισσότερο το παράρτημα. Εγώ θεωρούσα ότι από εκεί προκύπτουν όλα όσα είπα για την διαφάνεια. Αλλά καθώς υπάρχει και στην ιστοσελίδα, ίσως να μην χρειάζεται πράγματι. Σας παρακαλώ. Τσακ, τσακ. Αν θέλετε ιδιωτικέ συνομιλίε ενώ προσπαθώ να μιλήσω, παρακαλώ να βγείτε έξω. Ξέρω ότι έρχονται πολλοί τώρα για την ψηφοφορία, αλλά πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες ευπρεπίας. Είχαμε πει ότι δεν θα επισερχόμασταν σε θέματα νομοθεσίας ή πολιτικής, αλλά κυρίως διαδικαστικά θα το βλέπαμε. Ίσως όμως να είναι καλή ιδέα να συμπεριλάβουμε μερικές από τις ιδέες που είχαμε πει για τη διαφάνεια, όπου μερικοί εισηγητές φόρτωσαν όλα τα έγγραφα που είχαν λάβει στην ιστοσελίδα ως χρήσιμες πληροφορίες πέρα και από την απλή διαφάνεια. Γι' αυτό είχαμε θεωρήσει ότι την, στην επόμενη θητεία πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη τυποποίηση όλων αυτών. Για τις αποζημιώσεις με βάση αγορά κατάλαβα αυτά που είπες, αλλά εγώ τα λέω Excel approach. Ότι δηλαδή οι εταιρείες πατάνε σε αυγά, οπότε του ζητάνε να αποζημιώσουν. Αυτό ίσως είναι πιο πολύ θέμα νομοθεσίας και πολιτικής παρά διαδικασίας, αλλά τέλος πάντων. Ίσως να μπορούσαμε να οργανώσουμε κάποτε εν καιρό το τη μια ακρόαση, να βρούμε χρόνο να την κάνουμε, θα το κοιτάξουμε. Τέλος πάντων, περιμένω τις τροπολογίες. Η διορία λήγει 16 Δεκεμβρίου. Θα εξεταστούν τον Ιανουάριο στις 22 του μηνός και θα ψηφιστούν αργότερα τον Ιανουάριο. Μπορούμε όμως να πάρουμε και παράταση γιατί έχουμε χρόνο ως δική μας έκθεση. Πάει και αυτό λοιπόν. Και τώρα οι ανακοινώσεις της Προέδρου της Προέδρου που τις είχα βάλει για τώρα, αλλά έχω χάσει τα χαρτιά μου εδώ πέρα. Να τις, να Λοιπόν, πρώτον, γνωμοδοτήσεις και εκλισαβωνισμός ή λισαβονοποίηση πολλών οδηγιών και κανονισμών με αλλαγή των διαδικασιών σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Η οδηγία πολλές οδηγίες για τα στατιστικά ιδίως, για τις στατιστικές υπηρεσίες. Ο Γιώρη είναι υπεύθυνο και έχει πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου πρέπει να τα δει η νομική επιτροπή με συγχωρείτε είναι υπεύθυνη και θα ε, πρέπει να εξετάσει όλα τα θέματα ένα προς ένα. Μας ζήτησε η νομική επιτροπή να πληροφορήσουμε μάλλον ως επιστολή παρά ως επίσημη χρωμοδότηση, αλλά έτσι δεν θα υπάρχει επίσημη καταγεγραμμένη θέση της Οικονομικής Επιτροπής. Και γι' αυτό επειδή έχουν σημασία οι κατεξουσιοδότηση πράξεις για θέματα της εικόν, θα κάνουμε επίσημη γνωμοδότηση αλλά με επιταχυμένη διαδικασία μόνο στα αγγλικά. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι διανομή σήμερα, διορία τροπολογιών 4 Δεκεμβρίου στις 5, λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα, πάλι μόνο στα αγγλικά, και ψηφοφορία στις 9 Δεκεμβρίου στο Εστρασβούργο. Είναι ένα διαθεσμικό θέμα μεταξύ των οργάνων δηλαδή και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα έχετε καμία ιδιαίτερη δυσκολία με, τις με τη γνωμοδότησή μου. Αν παρέλειψα κάτι να μου το πείτε, αλλά συζήτηση παρετέρω δεν θα γίνει. Για τους επόμενους τριμερείς διαλόγους για το CFDR 28 Νοεμβρίου αρχίσαμε και είδαμε τα πρώτα μέτρα για το θέμα και παράλληλα τεχνική επεξεργασία, κυρώσεις, όροι λοιπά θα συνεχίσουν με γραπτή διαδικασία πριν τον επόμενο τριμερή διάλογο στις 8 Δεκεμβρίου. Ο ένατος τριμερής διάλογος για την Τραπεζική Ένωση άρχισε και υπάρχει συμφωνία για θέματα τρίτων χωρών και για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ενεργειακά. Η μόνη δυσκολία προς στιγμή είναι η κρατικές παρεμβάσεις όπου δεν σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος. Αύριο θα υπάρξει το τρίτο τριμερής διάλογος και στις 11 Δεκεμβρίου. Για τον τριμερή διάλογο κατάχρησης της αγοράς 28 Νοεμβρίου άρχισε και σημείωσε ιδιαίτερα το ρόλο της νομοθεσίας κλπ. ορισμό και καθορισμό του επίπεδου των κυρώσεων και δημοσίευση των συνεχίζει σε τεχνικό επίπεδο για ευθυγράμμιση με την οδηγία με τη σχετική οδηγία για την κατάχρηση των αγορών και τώρα κάτι που πρέπει να το ακούσετε πρέπει να γίνει επαναδιαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού για την τροποποίηση των οδηγιών 2003-71 και 2009 και λοιπά για, τη, για, τις για τις εξουσίες των ευρωπαϊκών οργάνων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και συμφωνίες για το ΣΚΑΡΠ που γενικά τα ονομάζουμε Omnibus, Omnibus 2 μάλιστα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Κακάρμπερτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ λίγα λόγια. Και η οδηγία Omnibus 2 για τη ρύθμιση της ασφαλής, του ασφαλιστικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί με το Omnibus 2 χωρίς προβλήματα. Ε, υπό τον Πίτερ Σκίνερ είχαμε το πρώτο κομμάτι για την αφαιρεγγιότητα, το οποίο συνεχίζει τώρα η Omnibus 2. Και στις δύο οδηγίες από την 1η Ιανουαρίου του 2016 αρχίζει η εφαρμογή. Και πιστεύω ότι με τη βελτίωση και τις αλλαγές που έχουμε φέρει με την Omnibus 2 μπορούμε και πάλι να ε, προωθήσουμε τα θέματα που είχε η ε, οδηγία για την αφαιρακαιοτητα ενα Ένα-δύο σημεία έχουν προς είχαν μείνει προς διευκρίνηση. Εν γέννη νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε καλές ικανοποιητικές λύσεις, ιδιαίτερα αποτελεσματικές και στην πράξη. Το σύνολο των μέτρων για τα μέτρα θα έχει πιστεύω σαν αποτέλεσμα ότι υπό δυσχερή συνθηκε στην αγορά και ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια ε, εφέτος θα επιτρέψει να προσφερθούν στους επενδυτές ιδιαίτερα ε, συμφέροντα πακέτα για επενδύσεις, επενδυτικά προϊόντα. Πιστεύω επίσης ότι η λύση στην οποία καταλήξαμε ήταν απαραίτητη, ήταν απαραίτητες. Και θέλω να ευχαριστήσω τους χειώδεις εισηγητές για την υποστήριξη που μου προσέφεραν και τη συνεργασία. Πάντα πολύ ευχάριστη, πάντα πολύ καλή. Για το Insolvency 2 και το Omnibus 2 ε, που ακολουθούν πιστεύω και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουν προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα, προστασία του καταναλωτή στις αγορές, τις ασφαλιστικές της Ευρώπης. Ήδη η Προεδρία του Συμβουλίου έχει προβλέψει ότι το Μάιο θα πάει στο Κορεπέρ. Εμείς τώρα πρέπει να περάσουμε το κείμενο από την επεξεργασία των γλωσσικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου. Αυτό θα μας πάρει κάποιο χρόνο. Καλό θα ήταν λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα αν μπορέσουμε να δούμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, το αργότερο του Μαρτίου, την Omnibus 2. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σβέν, θέλεις το λόγο. Συνήθως... Ε, δεν λαμβάνω το λόγο συνήθως για τέτοια θέματα, αλλά θα ήθελα εν συντομία να πω ότι δεν είδα ποτέ μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο να απέχει, να αποκλίνει τόσο πολύ και τόσο ριζικά από τις αρχικές του θέσεις. Και λοιπόν εν ώψη της ψηφοφορίας και με το τελικό αποτέλεσμα βλέπουμε σημαντική ελάφρυνση των προϋποθέσεων για την διασφάλιση, για τις ασφαλίσεις, οι μακροπρόθεσμες εγγύησεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι συνθήκες για την ε, δεύτερη οδηγία ε, για τι ασφαλίσει των παριθμών 2 του κύριου Σκίνερ. Τώρα έχουμε τις εγγύσει στα 67 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αποτελεί σε σημαντικό βαθμό αποδυνάμωση της προστασίας του ασφαλισμένου σε σχέση με τις αρχικές μας θέσεις. Επισημάνατε βέβαια και τις δυσκολίες της αγοράς. Πλην όμω, όσο αληθινέ και αν αυτέ οι δυσκολίε, τα μέτρα ε, στα οποία καταλήγεται δεν είναι η λογική συνέπεια της προσαρμογής της συνθήκης αγοράς. Αποτελούν μια καταγραφή των επιθυμιών των λόμπι, των μεγάλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έρχονται και εδώ για να ζητήσουν αυτό, διότι τελικά δεν έγινε δυνατό να διαμορφωθούν κοινέ και συνετικές θέσεις για την κοινή πολιτική και έτσι αφού ε, η Insolvency 2, η δεύτερη οδηγία για την αφαιρεγκαιότητα δεν έφερε τα αποτελέσματα που θέλανε, μεταφράστηκαν όσοι είχαν τα κείμενα που προτάθηκαν. Το Κοινοβούλιο λοιπόν όπως είπα έχει αποκλίνει όσο ποτέ άλλοτε από τις αρχικές του θέσεις. Δεν εξυπηρετείται η προστασία του καταναλωτή και κάθε ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα αξιοποιήσει με τις πιέσεις αυτές του Κοινοβουλίου την ελάφρυνση των απαιτήσεων για τις εγγύησει θα το πράξει. Θα δούμε στα επόμενα χρόνια ότι κάθε εταιρεία που αξιοποιεί αυτό το πλεονέκτημα εκτίθεται και στις πιέσεις αγοράς και οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν δυστυχώς ποιες είναι οι ασφαλιστικές εταιρείε που έχουν επαρκή αποθεματικά για να αντέξουν τις πιέσεις των ε, τιμών στην αγορά και ποιε είναι αυτές ε, οι οποίε θα του αφήσουμε στα κρύα του λουτρού. Αυτά είχα να πω. Ωραία. Από πλευρά σοσιαλιστών και δημοκρατών, ο Πίτερ Σκίνερ. Αυτή είναι μια νέα διαβούλευση της Επιτροπής. Ε, αν δώσουμε το λόγο στον ένα και ο λυπάμαι, πρέπει να δώσουμε και στους υπολείπους. Ο κύριος Σκίνερ. Ευχαριστώ. Πρέπει να λάβω το λόγο διότι το όνομά μου σχετίζεται με διάφορα ποσά, κυρίως εκατομμυρίων και ξέρετε ότι η θέση μου ήταν πάγια ευθύ εξ αρχής. Είμαι υπέρ ε, μιας εκ των υστέρων αξιολόγησης. Τελικά μια κάναμε ε, εκ των, υστέρων εκ των προτέρων συγγνώμη, και κάναμε εκ των αξιολόγηση και περιμέναμε και τα έγγραφα, ήρθαν τελευταία στιγμή και νομίζω ότι δεν έχουμε τα καλύτερα στοιχεία. έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι αξιοσημείωτα, δεδομένου ότι καθυστερήσαμε και πάρα πολύ να φτάσουμε ως εδώ. Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής είναι πάντα πιο σκληρές και τελικώς καταφέραμε ε, να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις με πιθανότητα να μην χρειαστεί να υποχωρήσουμε και σε τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν αξιοσημείωτη επιτυχία. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ήταν πολύ καλά. Καταφέραμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση με άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Ε, μέσω ε, μια διαδικασία στην οποία υποχρεώσαμε τι επιχειρήσει μα να τα πάνε πολύ καλά στον υπόλοιπο κόσμο και ε, πρέπει να υπάρχει και κάτι το ισοδύναμο από την άλλη πλευρά. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πολύ επιτυχής αυτή η διαπραγμάτευση και αυτό θα μα οδηγήσει σε παγκόσμιου κανόνε που θα οδεύουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Ε, να μπορούμε να αποφύγουμε συστημικούς κινδύνους, να περάσουμε σε πιο ισχυρά θεμέλια για τον ασφαλιστικό τομέα και αυτό μας χρειάστηκε 10 χρόνια. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και στους κοιόδης εισηγητές που συμμετείχαν με τόσο επικοδομητικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν εύκολος ο τελευταίος τριμερής διάλογος. Χρειάστηκε για 8 ώρες να προσπαθούμε να εμένουμε στις θέσεις μας. Και Πολλοί πίστευαν ότι δεν θα είχαμε καταφέρει να ε, πετύχουμε τίποτα και εμείς πέραν αυτού καταφέραμε να πετύχουμε και με ορισμένες διοργανικές αλλαγές και όλες αυτές ε, θα συμπεριληφθούν στην οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη ε, τα οποία θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει το λόγο διακαώς. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε ικανοποιημένοι πλέον μπορούμε να πάμε στο Omnibus 2 και μόλις ολοκληρωθεί θα ε, μπορέσει να περάσει από την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, τη δεύτερη του Φεβρουαρίου και ε, η ενυπόθηκη πίστη και σχετική οδηγία θα συζητηθεί πριν από το τέλος του 2013 και θα έχουμε και τις αλλαγές στον κανονισμό EPA που συμφωνήσαμε στο Omnibus 2. Ποιοι συμφωνούν υπέρ. Κατά. Σημειώνουμε λοιπόν ότι η πράσινη κατά. Έχουμε δύο ψήφους κατά. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε το σημείο της ημερήσιας διάταξης που μας περνάει στην ψηφοφορία. Να βρω ποιο νούμερο είναι. Λοιπόν, έτοιμοι. Ζαμπόλ, θέλεις το λόγο. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Βάλτε τις κάρτες σας, παρακαλώ. Πατήστε και τα κουμπάκια. Ωραία. Μία σύντομη ψηφοφορία έχουμε μόνο. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύσκολη είναι αυτή η αίθουσα για ψηφοφορία. Νομίζω ότι εγκρίνεται όμως. Συμβιβαστική τροπολογία Β σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ κατά. Να κάνουμε μια παλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα Προφορική τροπολογία α, αν δεν κάνω λάθος. Υπέρ. Κατά. Λυπάμαι. Είμαστε στην προφορική τροπολογία Α από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Προφορική τροπολογία Α. Ωραία. Απορρίπτεται. 16 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να κάνουμε μια παλήθευση όμως. Oops. I voted the wrong way. Oh well ψήφισα λάθος, αλλά τέλος πάντων και πάλι απορρίπτεται. Συγγνώμη. Ζητώ από την ομάδα μου. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω. Να κάνουμε μια ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 10. Θα προσπαθήσω να ψηφίσω σωστά αυτή τη φορά. Ζητώ συγγνώμη. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική τροπολογία C υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 40, 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση τη 45. No, that was rejected, sorry. Απορρίπτεται, ζητώ συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολο να δω ε, εδώ. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 17 γιατί δεν μπορούσα να δω ποιοι ψήφισαν τι Πέρασης εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά, ζητώ συγγνώμη. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία B από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ωραία να ψηφίσουμε Okay, um... Λοιπόν, Πρέπει να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε. Αυτό θα γίνει ηλεκτρονικά. «26 υπέρ, κανείς κατά και 11 αποχές». Να ψηφίσουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. closing the Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, καμία κατά και 11 αποχές. Δεν σκοπεύω να ψηφίσουμε την απόφαση για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, διότι χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία και δεν νομίζω ότι έχουμε απαρτία εδώ. Δεν θα αποφασίσουμε λοιπόν από αυτού σήμερα. Μπορούμε να το ξαναδούμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο, εάν έχουμε αρκετές παρουσίες. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία ε, για να μπορέσει να υπερψηφίσει η Επιτροπή. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Μπορεί και να το απορρίψουμε. Because Διότι ο συγητής δεν ζήτησε ακόμα την εντολή και επομένω, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Θα γίνει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Okay, Ωραία λοιπόν. Πέρασε τη συνέδρια σα.